Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Πριν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για τη δήλωση του Προέδρου Μπαρόζο μάλλον την παρουσίαση του, του Πρόεδρου Παρόζο για το πρόγραμμα εργασία τη Κομισιόν του 2011, θα ήθελα να θυμίσω ότι πριν 30 χρόνια έγινε ένα ε, φοβερό σεισμό που έπληξε κάποιε περιοχέ τη Ιταλία, την ε, Μπαζιλικάτα, όπου προκάλεσε χιλιάδε χιλιάδων θύματα. Πιστεύω πω όλοι μα μπορούμε να υπογραμμίσουμε την αλληλεγγύη μας προς τις οικογένειες όσο και προς τις περιοχές που επλήγησαν. Να δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο στον Πρόεδρο Μπαρόζο για την παρουσίαση του προγράμματος εργασίας ε, της Κομισιόν. Παρακαλώ κύριε Μπαρόζο, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα έχω την τιμή να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν για το 2011. Η παρουσίαση μπορεί να είναι η αρχή και το τέλος. Από τη μια πλευρά το πρόγραμμα ξεκινά μια νέα φάση πολύ σημαντικής πολιτικη εργασια Από την άλλη πλευρά η υιοθέτηση αυτού του προγράμματος αποτελεί το συμπέρασμα, την κατάληξη ενός ε, εντόνου διαλόγου ξεκίνησε εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο. Ε, η προετοιμασία αυτού του φετινού προγράμματος αποτέλεσε πρεμιέρα. Κατά την άποψή μου ήταν πολύ επιτυχής σε αυτή τη διαδικασία ε, Προχρονολογώντας ε, την ε, συμφωνία πλαίσιο, έχουμε ήδη θέσει προτεραιότητες για τα επόμενά, μας, ε, για τις, τα επόμενα χρόνια. Μέσω αυτής της νέας διαδικασίας σημειώθηκε μεγάλος βαθμός σύγκλησης σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίε. Είναι μια διαδικασία που στην ουσία παγιώνει αυτή την ειδική συνεργασία, όπως εγώ την αποκαλώ. Η ευρωπαϊκή δράση εστιάζεται σε αυτές τις προκλήσεις όπου μπορούμε να έχουμε απτή προστιθέμενη αξία. Οι 40 στρατηγικές πρωτοβουλίες τις οποίες ε, θέλουμε, θα ε, δεσμευόμαστε να παρουσιάσουμε το 2011 είναι πρωτοβουλίε οι οποίε έχουμε μαζί εντοπίσει και συμφωνήσει. Προ χάρη διαφάνεια θα περιλαμβάνονται και 150 άλλε προτάσει τι οποίε ε, εργάζεται, επί των οποίων εργάζεται η Κομισιόν. Βιώσιμη ανάπτυξη, εξασφάλιση τη ε, κοινωνική πρόνοια θα παραμείνει η προτεραιότητα για το 2011 και θα βασιστούμε σε τρει κύριου άξονα. Ενίσχυση τη διακυβέρνηση, ε, πλήρη μεταρρύθμιση του, του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώ και εφαρμογή της στρατηγικής 2020 για την ευφυή e e, βιώσιμη ανάπτυξη για όλους μέσω της έναρξης αυτού του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπως αποκαλείται, και την ε, ε, υποβολή των προτάσεών μας στις 29 Σεπτεμβρίου ενισχύουμε το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο και διευρύνουμε τη μακροοικονομική εποπτεία ώστε να εμποδίσουμε τις, ε, την έλλειψη ισορροπίας. Ε, έχουμε ήδη ξεκινήσει για μια σημαντική νομοθεσία η οποία έχει επιτευχθεί σχετικά. Το 2011 θα ολοκληρώσουμε τις νομοθεσίες, θα συντηρήσουμε τις προτεραιότητες όπως η διαφάνεια και θα εξετάσουμε την, ποιες ε, ε, ε, προτεραιότητες θα, προστα... θα, προωθήσουμε ώστε να αποφύγουμε μελλοντικές κρίσεις. Εμείς θα ζητήσουμε από το Συνοβούλιο και το Κοινοβούλιο να συμφωνήσουν για συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις το 2011. Θα πρέπει να εξακολουθήσουμε με τον ίδιο ρυθμό, να εστιάσουμε στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα στον 21ο αιώνα της παγκοσμιοποίησης. Και όταν οι ανταγωνιστές μας είναι φθηνότεροι, εμείς θα πρέπει να είμαστε ευφιέστεροι. Έχουμε αναπτύξει ως παράδειγμα πιο ανεπτυγμένο σύστημα ευρωπαϊκής τυποποίησης ως μια πλατφόρμα για την όξυνση της ε, ανταγωνιστικότητας των εταιριών μας, ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για να παραμείνει η ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξασφαλίσει περισσότερες και καλύτερες ε, θέσεις απασχόλησης, θα πρέπει να προγραμματίσει πολύ σωστά και προσεκτικά. Γι' αυτό η συγκέντρωση των πολιτικών, ε, κλιματικών αλλαγών, ενέργειας, μεταφορών και περιβάλλοντος θα είναι προτεραιότητα. Ιδιαίτερα ε, εστιάζουμε το 2011 στην ε, επάρκεια ενέργειας προσαρμοζόμενοι στη δυναμική οικονομική πραγματικότητα, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε προστασία των δικαιωμάτων εργαζομένων σε στενή συνεργασία με του κοινωνικού εταίρου. Και οι προτάσει κλειδιέ για την μετακίνηση εργαζομένων και για το χρόνο εργασία θα αναπτυχθούν μέσα στο 2011. Εν τω μεταξύ, η αναθεώρηση των, των κανόνων κρατικών ενισχύσεων θα είναι ένα απτό βήμα για τη θέσπιση ενό ποιοτικού πλαισίου που θα λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη φύση αυτών των υπηρεσιών με... Στην ε, νομοθεσία περί ενιαίας αγοράς έχουμε το φιλόδοξο στόχο να αποδώσει πλήρως η εσωτερική αγορά. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε σε επιχειρήσεις, όχι στη γραφειοκρατία και στις μικρόμεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά επιβαρύνονται πάρα πολύ και αποθαρρύνονται από το να ακολουθήσουν πολλά υποσχόμενα διασυνοριακά έργα. Ως συγκεκριμένο παράδειγμα, με το να ξεκαθαρίσουμε τους ε, κανόνες για το copyright και τη πνευματική διοκτησία που διαχειρίζονται συλλογικά θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και θέσεις εργασίας και διασυνοριακά, ιδίως στον πολλά υποσχόμενο ψηφιακό τομέα. Από την πλευρά της συζήτηση θα ενισχύσουμε κατά προτεραιότητα την εμπιστοσύνη των καταναλωτών με μια, ένα αναλλακτικό μηχανισμό επίλυσης ε, των διαφορών για να επιταχυνθεί αυτό το ζήτημα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είτε είμαστε φοιτητές, ταξιδιώτες, καταναλωτές ή οποιονδήποτε από τους άλλους πολλαπλούς ρόλους που έχουμε στην καθημερινή μας ζωή, όταν βλέπουμε τις νέες ευκαιρίες, ε, τις νέες εμπειρίες που έχουμε, όταν αυξάνεται η ποιότητα ζωής μας, τότε είναι η λογική η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στην υπηρεσία των πολιτών τη και το να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η πραγματικότητα για του πολίτε τη πρέπει να πηγαίνει πέρα από την ενιαία αγορά. Η ενίσχυση τη ασφάλεια θα πρέπει πάντα να έχει στόχο να βοηθήσει του πολίτε να αποφεληθούν από τι ευκαιρίε που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποτέ αυτός σκοπό. Η πρότασή μας για έξυπνα σύνορα θα διευκολύνει την ε, είσοδο και έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αποθαρρύνει την λαθρομετανάστευση. Επίση θα προσπαθήσουμε ε, και θα καταπολεμήσουμε αυτού που εκμεταλλεύονται για παράνομου σκοπού το οικονομικό μα ε, σύστημα και θα ανταποκριθούμε στι ανησυχίε των πολιτών στην εποχή του ίντερνετ. Η Ένωση πρέπει να παίζει ένα ρόλο στον κόσμο ανάλογο του οικονομικού, του οικονομικού της μεγέθους. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια συνοχή στις εξωτερικές μας δράσεις. Οπότε έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για τους στόχους 2020 ε, για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας διεθνώς επίσης για την αναπτυξιακή βοήθεια για, σε αυτούς στον κόσμο που χρειάζονται πραγματικά ισχυρότερη Ευρώπη. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, πριν να ολοκληρώσω, θα ήθελα να εξηγήσω λίγο το τι δεν θα βρείτε στο πρόγραμμα τη Κομισιόν και γιατί, όπω ανακοινώσαμε, θα υποβάλουμε προτάσει για το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο στα μέσα του 2011. Τα συγκεκριμένα μέσα και προγράμματα θα παρουσιαστούν το δεύτερο εξάμεινο του 2011 μαζί με το γενικότερο πλαίσιο για να διατηρήσουμε την πολιτική φύση του προγράμματος αυτού δεν έχουμε συμπεριλάβει τα της εφαρμογής. Το ίδιο και για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις καθώς βεβαίω το αποτέλεσμά της εξαρτάται από τρίτες χώρες. Βεβαίως οι δραστηριότητες αυτές είναι βασικό κομμάτι της δουλειά μας και θα συνεχίσουμε βεβαίως τον διάλογο μαζί σας επ' αυτών. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, Είπα στην εισαγωγή μου πως το πρόγραμμα εργασίας δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα του διαλόγου μας, αλλά και η αρχή της επόμενης φάσης των προσπαθειών μας για να βγει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την κρίση. Τώρα πρέπει να διατηρήσουμε την ορμή μας, να βρούμε τρόπους να επιταχύνουμε από κοινού το έργο μας. Οπότε θα ήθελα να ενθαρρύνω Κοινοβούλιο και Συμβούλιο να ε, έρθουν σε ένα τριμερή διάλογο για να δούμε πώ θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τι διατάξει για τον προγραμματισμό. Κατά την άποψή μα αυτό θα πρέπει να μεταφραστεί σε συμφωνίε για να οδηγηθούμε γρηγορότερα σε διαπραγματεύσει για κάποιε συγκεκριμένε πρωτοβουλίε ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Αυτό θα επιδείξει την αποφασιστικότητά μα για να έχουμε συγκεκριμένε έγκαιρε απαντήσει σε καιρού κρίσης που μας συγκλώνησαν όλου. Οι πολίτε τη Ευρώπη το αναμένουν αυτό και νομίζω πως τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανταποκριθούν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στους ε, ομιλητές εξ ονόματος των ομάδων, ξεκινώντας από τον ε, κύριο Ζώζεφ Σάιερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε Πιτέλα, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αξιότιμοι βουλευτέ. Πρέπει να ξεπεράσουμε την κρίση στην Ευρώπη, πρέπει να βασίσουμε την οικονομία μας στην εργασία. Τώρα αντιμετωπίζουμε μια σοβαρή κρίση και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να εξέλθουμε από αυτήν. Τι είναι το σημαντικότερο. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα εύρεσης εργασία όσο το δυνατόν περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες και θα πρέπει να υποστηρίξουμε στο πλαίσιο του προγράμματο εργασία τη δημιουργία θέσεων εργασία ω πολύ σημαντική προτεραιότητα. Έχουμε ξεκινήσει επίση μια επιταχυμένη διαδικασία για τη δημιουργία ενό νέου συστήματο οικονομική διακυβέρνηση και ελπίζουμε του χρόνου να έχουμε χρηματοοικονομικού κανόνε και νέε προτάσει για την οικονομική διακυβέρνηση και ελπίζουμε να υποβληθούν το συντομότερο δυνατόν για να τι εκρίνουμε και εμεί το συντομότερο δυνατόν. Υπάρχουν και κάποια άλλα μεμονωμένα ζητήματα, τα οποία εγώ θα ήθελα να θίξω, καινοτομία, έρευνα, ζωτική σημασία τομεί. Εδώ θα πρέπει να δούμε τι πρωτοβουλίες μπορούμε να αναλάβουμε. επίση πώ μπορούμε να προστατεύσουμε την πνευματική διοκτησία. Θα πρέπει να έχουμε και ένα ανταγωνιστικό σύστημα ευρεσιτεχνία στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό να αναπτύξουμε και τους ελέγχους των τροφίμων που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι περιμένουμε και από τους ίδιους παραγωγούς μας. Πρέπει να εφαρμοστούν κοινοί κανόνες. Επίσης θα θέλαμε να διατυπωθούν περισσότερες προτάσεις βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας. Να δούμε το νομοθετικό πρόγραμμα εργασίας, διότι ξεκινάει, ε, από τον Σεπτέμβριο ξεκίνησε, κάτι καινούριο. Το ανέφερε και στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης ο πρόεδρος ε, Μπαρόζο. Έχει σημαντικά προνόμια πλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να οδηγήσει στη λήψη επιπροσθέτων μέτρων. Δυστυχώς δεν ήταν καλή μέχρι τώρα η εμπειρία μας γιατί έχουμε δει μόνο ένα μέρος ε, του πρόγραμματος εργασίας να γίνεται πραγματικότητα και αυτό το έχουμε ε, πει και ξαναπεί. Χάνουμε ενέργεια, χάνουμε χρόνο για να αναλύουμε και να εγκρίνουμε έγγραφα κάθε χρόνο, ενώ τελικά αυτά τα έγγραφα, το περιεχόμενό τους στην πράξη δεν βλέπουμε να υλοποιείται. Κάθε χρόνο θα πρέπει να γίνεται μια αναθεώρηση, ίσως ακόμα και στη διάρκεια της χρονιάς θα πρέπει να γίνεται η ε, επισκόπηση, αξιολόγηση της πρόοδου των προγραμμάτων. Ευχαριστώ. Παρακαλώ όλους τους συναδέλφους να μένουν στα χρονικά όρια που τους έχουν δοθεί, γιατί ήδη με την προηγούμενη συζήτηση έχουμε ξεπεράσει το ωράριό μας. Σας παρακαλώ. Αυτό δεν το λέω επειδή πρέπει να μιλήσει ο κύριος Βόμποτα, ο οποίος πάντα είναι πολύ συγκεκριμένο και περιεπτικός. Θα προσπαθήσω. Κύριε Μπαρόσο, κύριε Αντιπρόεδρε, θεωρώ πως πολλά από τα πράγματα που αναφέρονται στο πρόγραμμα μας βρίσκουν σύμφωνους. Γι' αυτό θα ήθελα να αφαιρθώ περισσότερο στα κρίσιμα εκείνα σημεία κατά την απόψή μας. Βλέπουμε πως ε, η Ευρώπη επηρεάζεται όλο και περισσότερο από δυνάμεις αντιευρωπαϊκές ε, που μάχονται τα θεσμικά όργανα και πρέπει πραγματικά να σκεφτούμε ποιο περιεχόμενο και ποιες μεθόδους θα μπορέσουμε να αντιπαρατάξουμε σε αυτά. Πρώτα απ' όλα, η αναπτυξιακή πολιτική. Κύριε Πρόεδρε, καλά λέτε, πρέπει να ρυθμίσουμε τις χρηματαγορές, να έχουμε ομπρέλες κτλ. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτό το οποίο είχατε πει εσείς κύριε Πρόεδρε, αυτό το οποίο λέγαμε πράσινη ανάπτυξη κλπ. την αναδιάρθρωση της οικονομίας. Ο κύριος Έτιγκερ δημοσίευσε μια σειρά εγγράφων για την ενεργειακή πολιτική με τεράστιες επενδύσεις. Δεν μας λέει που θα βρει τα λεφτά πρέπει να βγούμε από την κρίση μέσω μιας πολιτικής ανάπτυξης. Και αναρωτιέμαι παραδείγματος χάρη στο τομέα τη ενέργεια, των συγκοινωνιών που θα πρέπει να γίνουν οι επενδύσεις, πώς θα γίνει για να δημιουργηθούν αυτές οι νέες θέσεις εργασίας. Δεύτερον, εσωτερική αγορά. Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να δημοσιευτεί αυτή η ε, έννοια της ε, εσωτερικής αγοράς και με παραπέμψετε στην έκθεση Μόντι, ο οποίος είχε κάποιες επικριτικές ε, διατυπώσεις για την κοινωνική διάσταση της εσωτερικής αγοράς. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα περισσότερα, γιατί θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και προς το συμφέρον των εργαζομένων, ότι δεν θα τους εκμεταλλευτούν για ντάμπινγκ μισθών. Τρίτον, φορολογική πολιτική. Το είδαμε ήδη και στο παράδειγμα με την Ιρλανδία πως δεν είναι δυνατόν κάποιες χώρες να έχουν χαμηλότερους φόρους για να προσελκύουν επιχειρήσεις και μετά όταν έχουν οικονομικές δυσκολίες να πούνε σε άλλες χώρες «Ε, κοιτάξτε βοηθήστε μας με τον προπολογισμό γιατί έχει ελλείμματα. Η φορολογική εναρμόνιση ως ένα βαθμό όπως παραδείγματο χάρη με ελάχιστα ποσοστά φόρων στις επιχείρησεις είναι απολύτως απαραίτητη. Ξέρω πως δυσκολεύεστε πάρα πολύ να πείστε τα κράτη-μέλη, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης για τον κοινωνικό τομέα τα ανέφερα, η ψαλίδα μεταξύ πλουσίων και φτωχών είναι απαράδεκτη. Πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα τα της στόχες. Και τέλος, μιλήσατε για τις ανησυχίες των πολιτών. Πράγματι είναι πολύ σημαντικό, αλλά και το πώ λέμε και το πώς παρουσιάζουμε αυτά τα οποία κάνουμε εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έχουμε κάτι τι ανάγνωσε ανακοινώσει τύπου πρέπει να παρουσιάσουμε καλύτερα την δουλειά μας. Παραδείγματο χάρη με τις πρωτοβουλίες ε, πολιτών. Αν χρησιμοποιηθεί αυτό από αντιευρωπαίους, Εμεί θα πρέπει να βοηθήσουμε να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπου που είναι υπέρ τη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντίνα Ζωάνα Βαλεάν για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε Μπαρός, αγαπητοί συνάδελφοι. Η καιρή είναι δύσκολη για την ευρωπαϊκή οικονομία και για το ευρωπαϊκό σχέδιο γενικότερα. Έχουμε μιλήσει για μεγάλες στρατηγικές όπως το κλιματικό πακέτο, στη στρατηγική 2020, προγράμματα επί προγραμμάτων, ωστόσο δεν φαίνεται να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε και ποιοι θέλουμε να είμαστε. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί το να θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι δεν αρκεί για να είμαστε όντως οι καλύτεροι, ενώ είμαστε μπερδεμένοι σε στρατηγικές, δεν πιστεύουμε όλες αυτές. Κανείς ή σχεδόν κανείς δεν τις εφαρμόζει και κανένας δεν είναι έτοιμος να τις χρηματοδοτήσει. Φαίνεται να έχουμε ένα σωρό στρατηγικές, ενώ δεν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον να υλοποιηθούν. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε οι βάσει, τα βασικά στοιχεία που έφτιαξαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και μα συγκέντρωσαν όλου μαζί. Τα απλά φυσιολογικά πράγματα. Η νέα χώρα θα πρέπει να είναι το μεγάλο μα πρόγραμμα και να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να την επιβάλλουμε. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, θα χρειαζόμαστε περισσότερη οικονομική ολοκλήρωση και ο μόνο λογικό τρόπο για να γίνει κάτι τέτοιο είναι η νέα αγορά. Εγώ καλωσορίζω το πρόγραμμα εργασία τη Κομισιόν και ιδιαίτερα την πρότασή σα για το Ινενιά αγορά, αλλά δεν είναι αρκό. Ξέρετε, έχετε την έκθεση Μόντι, ξέρετε τι χρειάζεται, να ενθαρρυνθούν οι επενδύσει, να προσερκίσουμε το κεφάλαιο, να περικόψουμε τι γραφειοκρατικέ δαπάνε, ε, απλά πράγματα που έχουν επιρροή για την ανταγωνιστικότητα, ε, περιορισμό των ενεργειακού κόστο, μεταρρύθμιση τη γεωργική πολιτική, το μέλλον των μεταφορών, η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο πρέπει να δουλεύουν και ε, ε, συντονισμένα Γι' αυτό προσβλέπουμε σε ένα φιλόδοξο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μέσα στο 2011. Τώρα, χρειάζονται περισσότεροι κανονισμοί για να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση, ναι, αλλά αν ο στόχος είναι το να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Πάντως, θα πρέπει να αποφύγουμε να υιοθετήσουμε μια αυτιστική απάντηση στην κρίση, ελπίζοντα ότι ο υπόλοιπο κόσμος θα ακολουθήσει. Η Ένωση δεν είναι μια ένωση ιδεών, κεφαλαίων και αξιών, δεν, είμαστε, δεν θα είμαστε ο παγκόσμιο παίκτη που θέλουμε να είμαστε και αντί να επηρεάζουμε τι πολιτικέ του κόσμου, θα επηρεαζόμαστε εμεί από αυτέ. Και τώρα δύο λόγια για το Ευρωπαϊκό Εξάμενο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε καλύτερη θέση για να εντοπίσει ε, τα ισχυρά και τα δύνατά μα στοιχεία όταν προγραμματίζει τη δουλειά τη. Αλλά προσέξτε, γιατί αυτό που προτείνεται στου πολίτε και στα κράτη-μέλη να πιστεύουν ότι οι Βρυξέλλε τα ξέρουν καλύτερα ότι η πολιτική των Βρυξελών είναι πιο κοντά στους συμφέροντα των πολιτών και πιο κοντά στις περιφέρειες τους. Είναι δύσκολη δουλειά και δεσμεύεστε σε αυτό μέσω του συντονισμού των πολιτικών για το 2011. Εύχομαι ότι θα καταφέρετε να το αποδείξετε, ότι θα προωθήσετε τις δουλειές, τις θέσεις απασχόλησης και την ανάπτυξη όχι για κάποιους αλλά για όλους, γιατί διαφορετικά ο πραγματικός αντιευρωπαϊσμός θα αυξηθεί. Σας εύχομαι καλή τύχη. Ευχαριστούμε συνάδελφο. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Ρεμπέκα Χάρμς για τρία λεπτά. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπαρόζο. Σημαντικό είναι να ξεκαθαρίσουμε πως δεν μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το πρόγραμμα εργασίας χωρίς να αναφερθούμε στα όσα συμβαίνουν στον προπολογισμό αυτή τη στιγμή. Χωρίς να αναφερθούμε στο θέμα Ελλάδα-Ιρλανδία και πιθανώς και άλλες χώρες που θα αντιμετωπίσουν προβλήματα. Θα ήθελα να πω αυτό το οποίο άκουσα στο κλείσιμο της συζήτησης ε, του προπολογισμού, πως ε, είσαστε ανοιχτό στη θέση του Κοινοβουλίου και αυτό είναι πραγματικά σημαντικό. Δηλαδή να είμαστε ειλικρινεί για το πρόγραμμα αυτό της εργασίας. Μην παριστάνουμε δηλαδή ότι μπορούμε να επιτύχουμε όλους αυτούς τους στόχους αν δεν έχουμε έναν ανάλογο αξιόπιστο προϋπολογισμό που δεν θα αποτελεί αντικείμενο διαφωνίας κάθε χρόνο. Δεύτερον, θεωρώ πως η συζήτηση περί Ιρλανδίας κατέδειξε σε ποιο βαθμό είμαστε μακριά από μια πραγματική λύση και διέξοδο από την κρίση. Κρίση στην οποία βρεθήκαμε γιατί ήμασταν πολύ φιλελεύθεροι όσον αφορά τις χρηματαγορές και για την ομάδα μου θα ήθελα να πω πως αυτό το οποίο υποβάλλατε από πλευράς προτάσεων για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την ε, οικονομική κρίση και τις διεξόδους. Υπάρχουν κάποια καλά σημεία εκεί πέρα, αλλά δεν θεωρούμε πως ο στόχος τον οποίον έχετε θέσει επαρκεί Και αν δούμε ήδη πόσο καιρό συζητάμε και λέμε πόσο επιτυχημένη είναι η νομισματική μας ένωση, αν θέλουμε πραγματικά να το εγγυηθούμε, θα πρέπει να πάμε σε αυτή την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης. Δεν γίνεται αλλιώς. Οπότε να βγούμε θετικά από την κρίση σε περισσότερη κοινή οικονομική πολιτική. Να μην αντιμετωπίζουμε μόνο το σύμπτωμα. Αυτό λείπει από την πρότασή σας και αυτό θα δούμε. Ο κύριος Φοποντα ανέφερε ήδη τα πράσινα θέματα. Πρέπει να πω πως δεν είμαι ικανοποιημένη με το πώς ε, αυτό το οποίο περιγράφεται στρατηγική 2020 ως αηφόρος ε, και δίκαιη ανάπτυξη το πώς μεταφράστηκε στο πρόγραμμα εργασίας. Ε, δεν είναι αυτό, αυτό το οποίο είχαμε πει περί Ευρώπης 2020. Ο κύριος Έτιγκερ είναι ένας από τους επιτρόπους που πάντα κινείται μακριά από την ιδέα της ευρωπαϊκής αηφορίας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Βλάσεκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, το 2012 ε, θα είναι ένα έτος ε, δοκιμής ε, για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την οικονομική ανάκαμψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εξού και το πρόγραμμα για ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε αυτό το πλαίσιο θέλω να πω ότι κάποιες φορές ε, η λιγότερη νομοθεσία ε, σημαίνει περισσότερα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε με κάποια ανησυχία κάποιες από τις ρυθμιστικές δραστηριότητες. Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι Υπάρχουν ε, ε, κάποιες ε, υποθέσεις στο δικαστήριο που συνηγορούν υπέρ της μία έκδοσης αδειών σε κάποιους τομείς. Και πραγματικά υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες θα πρέπει στη φάση της υλοποίησης, στη φάση της εκτέλεσης επίσης να είναι όλοι έτοιμοι για την ε, προετοιμασία. Κυρία Λεϊαρίκ, για ανάμεση. Ο κύριος Λεϊαρίκ, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε Μπαρόζο, φαίνεται ε, η Επιτροπή να μην έχει υπόψη της τη σοβαρή κρίση που βιώνει η Ευρώπη. Στο έγγραφό σας μάλιστα λέτε ότι είναι ξεκάθαρα τα σημάδια της ανάκαμψης. Πού τα βλέπετε για τους φτωχούς, για τους αστέγους, ε, για τους ανέργους. Ξέρετε ότι πάνω από 400 δις δημόσιου χρήματος ε, δίνονται για να στηριχθούν σήμερα οι τράπεζες και ξέρετε ότι ακριβώς αυτά τα 400 δις ε, οικονομιών επιβλήθηκαν στις 8 χώρες, στους πολίτες των 8 χωρών που είναι σε σχέδια λιτότητας, άρα το πρόγραμμά σας είναι αναποτελεσματικό. Σας προτείνω λοιπόν προβείται προβείτε σε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για του εργαζομένου και τους Ευρωπαίους πολίτες ό,τι αφορά την υλοποίηση των συνθήκων ε, του Μαστρέχτ και της Λισαβόνας. Γιατί δεν νομίζω ότι η λύση είναι η δημοσιονομική ε, λιτότητα, η μισθολογική λιτότητα, αλλά αντίθετα αύξηση τη αμοιβή τη εργασία, βελτίωση τη κοινωνική προστασία και των συνταξιδοτικών συστημάτων, μια αλληλέγγυα ανακατανομή. Θα πρέπει ε, να υπάρξει δίκαιη κατανομή των κεφαλαιοχικών εισοδημάτων, φορολογική δικαιοσύνη και γιατί να να μην ξεκινήσει άμεσα μία μελέτη για την φορολόγηση των κινήσεων κεφαλαίου. Επίσης ένας νέος ρόλος για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ένα ε, κονδύλι που θα βοηθήσει τα κράτη να χρηματοδοτήσουν τι τράπεζε για την εξασφάλιση τη εργασία, για την κατάρτιση, την εκπαίδευση, για όλα τα δημόσια αγαθά με τι νέε δημόσιε υπηρεσίε ε, καινοτομία και έρευνα. Σήμερα μιλάμε για ανακατανομή και αναδιανομή του πλούτου. Δεν θα πρέπει να κλείσουμε τον κόσμο στο κλειό τη ανεργία ε, και τη λιτότητα. Σα ευχαριστούμε κύριε Λαγιαρίκη. τώρα η κυρία Νίκη Τζαβέλα για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αφού η δημιουργία των θέσεων είναι προτεραιότητα του προγράμματος, εγώ θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της Κομισιόν, αλλά φοβούμαι πως αυτή τη στιγμή δεν με ακούει κανείς από την Κομισιόν. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της Κομισιόν και πάλι, κύριε Πρόεδρε, σε μια νέα περίοδο μετανάστευσης που γίνεται από την βότια Ευρώπη προς τα έξω. Ήδη στην Ελλάδα βλέπουμε τεράστιους αριθμούς νέων που φεύγουν για την, Αυστρία, την, την Αυστραλία, συγγνώμη, τον Καναδά και τα Εμμυράτα. Το ίδιο γίνεται και στην Ιρλανδία. Από την άλλη πλευρά η Γερμανία ανακοινώνει ότι έχει έλλειψη δικευμένου εργατικού δυναμικού. Αυτό που λέμε τώρα είναι ότι η Γερμανία δεν χρειάζεται να εισάγει ειδικευμένο εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Χώρες κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα θα μπορούσαν να δώσουν ειδικευμένο εργατικό δυναμικό στη Γερμανία. Εγώ θα ήθελα να προτείνω με μια πρωτοβουλία για την Κομισιόν. Προχωράτε με την έννοια της προστεθέμενης αξίας. Γιατί δεν υιοθετείτε μια αγορά εργασίας ευρωπαϊκής προστεθέμενης αξίας. Το θέμα πως τα κράτη-μέλη πρέπει να καλύψουμε την ε, ζήτηση και την ε, παροχή να δώσουμε στην Ευρώπη ε, ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Λείπει αυτό από το πρόγραμμα και το προτείνω. Σας ευχαριστούμε. Το λόγο έχουν τώρα οι ομιλητές που έχουν εγγραφεί για τη συζήτηση. Ξεκινάμε με τον κύριο Ρίτσαρντ Σίμπερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την Κομισιόν για το φιλόδοξο πρόγραμμα εργασία, αλλά νομίζω πως θα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στους στρατηγικούς στόχους της Ένωσης και θα πρέπει να κοιτάξει πιο θαραλέα και χωρίς φόβο η Κομισιόν στο μέλλον. Βεβαίω, εδώ πέρα το Συμβούλιο φρενάρει και οι προοδευτικέ δυνάμεις θα πρέπει να διατηρήσουν ένα κοινό μέτωπο. Η ανταγωνιστικότητα είναι κεντρικό σημείο. Πρέπει να παραμείνει η ανταγωνιστική Ευρώπη για να επιτύχουμε τους στόχους μας της ε, αηφόρου και κοινωνικής ανάπτυξης. Σημαντικό είναι βεβαίως το πώ θα πουλήσουμε, αν θέλετε, αυτό το μήνυμα. η δυνάμεις οι εχθρικές προς την Ευρώπη είναι πολύ παρούσες στα ΜΜΕ, όλοι ε, όμως γνωρίζουν πως η Ευρώπη μόνο από κοινού μπορεί να πάει προς σωστή κατεύθυνση. Συνολικά νομίζω πως θα πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν να βάλει στο πρόγραμμά της τον τίτλο «Αύξηση της αποτελεσματικότητας». Είτε μιλάμε για τους πόρους, την ενέργεια, αλλά στην εκπαίδευση, στα πανεπιστήμια παντού πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεισφορά για τη δημιουργία της έξυπνης Ευρώπης και εδώ πέρα ειδικά στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης απαιτούνται προσπάθειες. Δεν κοιμάται ο υπόλοιπος κόσμος, αλλά βεβαίως αυτό δεν σημαίνει πως θα πρέπει να κοιτάμε φοβισμένοι το μέλλον και να ασκούμε την πολιτική που κάνει το Συμβούλιο έτσι, του μικρό κρατικού συμφέροντος. Ευχαριστώ για δύο λεπτά. Έχει το λόγο η κυρία Μόνικα Μπενόβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πως ε, στους ταραγμένους αυτούς καιρούς δεν ήταν βεβαίως ε, εύκολο για την Κομισιόν να υποβάλει ένα τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα, γι' αυτό σας συγχαίρω. Λέξη κλειδί βεβαίως εδώ πέρα είναι η ανάκαμψη και η αηφόρος ε, ανάπτυξη. Είμαι όμως κάπως επιφυλακτική. Είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλήσουμε για ανάκαμψη. Υπάρχουν κάποια σημάδια, αλλά δεν είναι σίγουρο πως ε, μπορούμε να μιλήσουμε για ανάκαμψη. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε άλλες τέτοιες ε, περιπτώσεις ε, σαν αυτές τις οποίες είχαμε. Βλέπουμε πως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία. Τα χρέη είναι πάρα πολύ μεγάλα, αλλά με τις περιεριστικές πολιτικές μόνο μεγαλύτερα θα γίνουν παρόμοια είναι η κατάσταση και ε, με την ε, επιβολή αυστηρότερων κανόνων για τον προπολογισμό. Είναι αντιπαραγωγικά αυτή τη στιγμή. Η πειθαρχία στον ε, προϋπολογισμό δεν αντιμετωπίζει την διαρθρωτική ανισορροπία στην Ευρώπη. Αυτό είναι θέμα βεβαίως μιας άλλης συζήτησης. Υποστηρίζω επίσης την ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Δεν ξέρω αν επαρκούν τα μέσα τα οποία προτείνονται, αλλά κατά βάση μιλάμε για ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Μια προσπάθεια για η ανάπτυξη επίσης είναι θετική και αντιλαμβάνομαι πως το πρόγραμμα αυτό βέβαια δεν μπορεί να πάει σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά πρέπει να καταπολεμηθεί και η φτώχεια και να έχουμε πιο φιλόδοξο πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης. Σας ευχαριστώ κυρία Μπένοβα και επειδή τελειώσατε με ένα δευτερόλεπτο λιγότερο χρόνο από ό,τι σας είχαμε δώσει. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Χάτουν για ένα λεπτό. Το πρόγραμμα της Κομισιόν συμπεριλαμβάνει κάποιες αξιόλογες προτεραιότητες, η βιώσιμη ανάπτυξη, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην ενέργεια, πρόθεση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ε, ε, είναι εμείς είμαστε υπέρ όλων αυτών των ε, φιλοδοξιών και ελπίζουμε πως όντως θα επιτευχθεί η πρόοδος και για άλλες προκλήσεις, όχι μόνο για αυτές. Η, ομάδα Ευρωπαϊκή Συμμαχία που συμπεριλαμβάνεται SNP αλλά και άλλους ε, Ευρωπαίους εθνικιστές από την ε, Ουαλία, την Καταλωνία και την Φλάνδρα ε, είναι, φιλοδοξούν να παίξουν ρόλο στην λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνοντας ε, ε, μέρος ως ανεξάρτητα κράτη-μέλη ώστε να μπορούμε επικοδομητικά εδώ να λειτουργήσουμε ως συνάδελφοι για μια καλύτερη Ευρώπη. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Βέραντελ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή κρίσης που βιώνουμε υπάρχουν δύο μεγάλα είδη πολιτικής και δράσεων. Πολιτικές και δράσεις προληπτικού χαρακτήρα και πολιτικές και δράσεις ε, όθησης. Οι πρώτες είναι αυτές τις οποίες πρέπει να φέρουμε σήμερα σε πέρας με την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με την ε, διακυβέρνηση και την ενίσχυσή της και ό,τι άλλο θα μας προειδοποιεί για το ότι υπάρχουν προβλήματα πριν ξεχυλήσουν ε, και δημιουργήσουν πρόβλημα για τις ε, ευρωπαϊκές οικοδομίες αυτά τα προβλήματα. Το δεύτερο είδος όμως πολιτικών, ε, όθησης δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι πολιτικές. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εκπρόσωποι της Επιτροπής που είστε παρόντες, ε, θέλω να σας πω το εξής. Αυτές οι πολιτικές όθησης υπάρχουν τρεις βασικές πτυχές φυσικά, πολλέ, αλλά εγώ τρεις θα αναφέρω μόνο. Έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη ψηφιακή ε, και εσωτερική αγορά. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, ε, την έρευνα και την καινοτομία, εκεί εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν ελλείψεις στο πρόγραμμα εργασία το οποίο μα παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έλεγε πριν ο πρόεδρο Μπαρόσο ότι θα έλθουν και τα ειδικά προγράμματα στα μέσα του 2011. Εγώ νομίζω όμω ότι αυτό δεν αρκεί σε μένα και στην ομάδα μου θα μας άρεσε περισσότερο να έχουμε ήδη τώρα μνήα ε, στο, πρόγραμμα, στο 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Δεν υπάρχει τέτοια μνήα στην πρόταση όμως της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Βιζονέν για ε, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι τυπική διαδικασία, είναι ένας, στόχος να προσελκύσουμε την, ένας τρόπος να προσελκύσουμε την προσοχή των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και ένας τρόπος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει μια ιδέα για τους τομείς ε, από τους οποίους, στους οποίους μπορεί να αναμένει την υποστήριξη των Ευρωβουλευτών. Θα είναι σημαντικό να δούμε τι κάνει η Ευρώπη του χρόνου σε διεθνές επίπεδο, στο διεθνή στίβο. Θέλουμε μια ισχυρή υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Αυτό θα είναι σημαντικό και πρέπει να το λάβει υπόψη η Επιτροπή στο πρόγραμμα εργασίας της. Θα ήθελα επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει και να επεξεργαστεί και τα περί διεύνησης, όπως έκανε το 2010. Το κεφάλαιο 23 πολύ σημαντικό. Και ελπίζουμε στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κάνει μια αναφορά σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις. Επίσης, ό,τι αφορά την Τουρκία, που είναι σημαντικό και αυτό, πρέπει οι δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί να τηρηθούν και θα πρέπει ε, η τουρκική πλευρά βέβαια να συνεχίσει και τις προσπάθειες για το Σύνταγμα, το νέο Σύνταγμα και για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα θέλαμε επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώνει σε τακτά διαστήματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά και την αίτηση της Σερβίας. Ελπίζουμε η πολιτική γειτονία να οδηγήσει στις απαιτούμενες διορθώσεις ώστε να υπάρξει συντονισμός μεταξύ αφενός των στόχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφετέρου του προπολογισμού για την επίτευξη αυτών των στόχων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια είναι έτοιμο να υποστηρίξει τη στρατηγική για το 2020. Ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Ανδρέας Σβάμπ για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι. Εμείς θέλουμε το νομοθετικό πρόγραμμα της Κομισιόν να προσανατολίζεται στους μακροπρόθεσμους στόχους και πρέπει άρα να βελτιωθεί κάπως. Αν και βεβαίως συμφωνούμε στα βασικά. Στον τομέα της εσωτερικής αγοράς ήθελα να πω πως ε, αν θέλουμε να επιτύχουμε αυτά τα οποία λέει ο κύριος Μόντι θα πρέπει όλοι οι πολίτε τη Ευρώπη να υποφεληθούν από αυτήν την εσωτερική αγορά και ακόμη περισσότερο αν θέλετε. Εάν δούμε λοιπόν το πρόγραμμα εργασίας της ε, Κομισιόν, αυτό σημαίνει πως πρώτα απ' όλα η Κομισιόν θα πρέπει να ενισχύσει τις διαδικασίες επί παραβάση κατά των ε, κρατών μελών ειδικά και στι περιπτώσει υπέρβαση του ελλείμματο. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο εδώ μέσα. Επίσης, αυτά τα οποία αφέρθηκαν, ε, στεγαστική πίστη, ψηφιακή ατζέντα, πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν συζητήθηκαν, τα οποία χρειαζόμαστε μα περιπτώσει έτσι ώστε τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί για το 2011 να υποβληθούν από τώρα. Δεν μας βοηθάει βεβαίως πάρα πολύ εδώ η Κομισιόν. Και το τελευταίο το οποίο θα ζητούσα από την Κομισιόν είναι όλες οι νομοθετικές προτάσεις να έχουν μία αξιολόγηση αντικτύπου για να δούμε αν είναι αναγκαίες. Ευχαριστώ κύριε Σφάμπ. Τώρα τον λόγο έχει η κυρία Εύελιν Γκέπχαρτ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Θεωρώ πως με τη συνθήκη της Λισαβόνας κάναμε ένα μεγάλο βήμα για τους πολίτες μας καθώς ε, εισήχθη έτσι η κοινωνική οικονομία της αγοράς στις αρχές της ευρωπαϊκής πολιτικής και είναι σαφές πως ως Ευρωπαίοι, ως βουλευτές αναμένουμε η κοινωνική οικονομία της αγοράς να μεταφραστεί σε κάτι πραγματικό. Και τώρα βλέπουμε τι περιέχει η νομοθεσία αγοράς και λείπουν εκεί πέρα κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν. Δεν επαρκεί να γίνει μια μελέτη κοινωνικού αντικτύπου. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι μια κοινωνική ρήτρα, έτσι ώστε αυτό το οποίο μας έχουν υποσχεθεί, δηλαδή ότι και οι πολίτες θα έχουν όφελος από την Ευρώπη, να μπορούμε να το δούμε και να μην είναι μόνο στα χαρτιά. Και το θέμα δεν είναι μόνο η κοινωνική ρήτρα. Είναι τόσο σημαντικά πράγματα όπως παραδείγματος χάρη οι υπηρεσίες κοινή ωφελία που χρειάζονται ειδική προστασία και δεν βλέπω εδώ πέρα την Κομισιόν να ασχολείται με αυτό το θέμα ή το ζήτημα των εργαζομένων κάπως πιο έντενα στην ε, οδηγία περί απόσπασης. Οπότε έχω εξοργιστεί εδώ και καιρό απαιτούμε ως Κοινοβούλιο από την Κομισιόν να δημιουργηθεί επιτέλους ένα σύστημα μαζικών προσφυγών. Υπάρχουν 6-7 διαφορετικές μελέτες της Κομισιόν και τι διαβάζουμε εδώ πέρα στο πρόγραμμα της Κομισιόν, άλλη μία μελέτη. Ε, δεν γίνεται θέλουμε επιτέλους προτάσεις και αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Γκέπχαρτ. Ο λόγο ο κύριος ε, Ζαν Πολ για να μην λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ω συντονιστή του ΕΛΚ στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, ε, θέλω να επιμείνω σε δύο σημεία του προγράμματό σα. Πρώτα απ' όλα, ενίσχυση τη οικονομική διακυβέρνηση έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Υποδεχθήκαμε με ικανοποίηση το πακέτο για την οικονομική διακυβέρνηση. Η επιτεύξη του στόχου αυτού είναι πρωταρχική σημασία και σε αυτό το τομέα θέλουμε ε, αποτελεσματικά και δεσμευτικά μέτρα στη δική μα ομάδα, τα οποία να υπερβαίνουν τα προτινόμενα μέτρα. Επίση, αναγκαίο είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει πραγματικά στην ε, υλοποίηση ε, και την εφαρμογή των διαφόρων πολιτικών και μέτρων. Θα πρέπει να βρεθεί μια νομική βάση για να μην ε, χρειαστεί ε, σημαντική τροποποίηση των συνθήκων που θα καθυστερήσει την εφαρμογή των μέτρων που είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν. Το δεύτερο σημείο είναι η συνέχιση των δράσεων σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά. Έχουμε προτάσεις επιτάπητος θα υλοποιηθούν είναι αποφασιστική σημασία στο έτος 2011. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ δείχνει θέληση. Το 2010 και το Κοινοβούλιο έδειξε τη θέλησή του για την υλοποίηση, του, για την υιοθέτηση μάλλον του πακέτου για την εποπτεία και θα πρέπει και να έχουμε και τον κανονισμό για την ευρωπαϊκή εποπτεία ε, των οίκων αξιολόγηση μέχρι τα τέλη του έτους. Θέλουμε να συνεχίσουμε ε, στην κατεύθυνση πραγματικών ε, φιών νομοθετημάτων που θα έχουν αποτελεσματικότητα. Αυτό άλλωστε περιμένουμε σήμερα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκοζέ. Ο κύριος Ντερόσα για 1,5 λεπτό έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ο πρόεδρος Μπαρόσο μίλησε στην εισαγωγή του για τη θέσπιση μέτρων σε ό,τι αφορά την απόσπαση των εργαζομένων, αλλά δεν ήταν ξεκάθαρο, δεν ήταν πολύ συγκεκριμένο. Πάντω, ανέλαβε μια συγκεκριμένη δέσμευση στι ακροάσει ε, που προηγήθηκαν ε, του ορισμού του. Μίλησε ότι θα υπάρξει αναθεώρηση οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων για να μην υπάρχει κοινωνικό dumping και ξέρουμε για κάποιες πολύ σημαντικές υποθέσεις και προβλήματα που υπήρξαν. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εισαχθεί νομοθεσία η οποία θα παρέχει ασφάλεια δικαίου για αυτούς τα κράτη-μέλη που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίε γενικού ενδιαφέροντος. Φαίνεται να υπάρχει πλήρη τύφλωση ε, της Επιτροπής ε, απέναντι στο πρόβλημα αυτό. Εγώ επεξεργάζομαι μια έκθεση και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό στις αρχές ίσως του επόμενου έτους. Θα πρέπει να πω επίσης ότι μου αρέσει πολύ και η πλατφόρμα για τη φτώχεια, αλλά δεν έχω καμία ένδειξη για το ότι η Κομισιόν χρησιμοποιεί τη στρατηγική 2020 στην οποία βασίζεται η πλατφόρμα, παραδείγματο χάρη στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις με την Ιρλανδική κυβέρνηση για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα. Αν η στρατηγική 2020 δεν είναι το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, τότε ποιο είναι το πλαίσιο. Ποια είναι η ευρωπαϊκή συμμετοχή, συνεισφορά στην επίλυση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Ιρλανδία πέραν της διάσωσης τραπεζών. Ένα τελευταίο σημείο μου επιτρέπετε. Νομίζω ότι βάζουμε, ε, προτρέχουμε. Έχουμε τον εταιρικό φόρο, αλλά δεν μιλάμε για κοινή φορολογική πολιτική. Δεν έχουμε έναν προπολογισμό επαρκή για τις ε, περιφερειακές ε, χώρες, τις απόκεντρες χώρες. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια τέτοια ευρωπαϊκή πολιτική και μετά να μιλήσουμε για τον εταιρικό φόρο που θα είναι και ο ίδιος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λόγο έχει ο κύριος Όρη για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ είμαι συντονιστή του ΕΛΚ για, στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και καλωσορίζω το πρόγραμμα εργασίας καθώς και το γεγονός ότι μπορέσαμε να μιλήσουμε για την πρωτοβουλία για τις νέες θέσεις απασχόλησης. Εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιες πολιτικής φύσης παρατηρήσεις. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να φτάσουμε σε συμφωνία και η Κομισιόν να μην εξετάζει μόνο τα όσα προτείνει το Συμβούλιο αλλά να λάβει πλήρως υπόψη τις προτάσεις και το χρονοδιάγραμμα που προτείνει το Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό και πολλοί προηγούμενοι ομιλητέ το ανέφεραν. Θα πρέπει να έχουμε αποθεματικά για τον προπολογισμό, για τα προγράμματά μα και τι προτεραιότητέ μα και προσδίδω μεγάλη σημασία ταυτόχρονα στο γεγονό ότι τα καθορισμένα προγράμματα να είναι προγράμματα που μπορούν να μετρηθούν και να παρακολουθηθούν. Επίση, μιλάμε για βελτίωση του επίπεδου εκπαίδευση και κατάρτιση. Ωστόσο, αυτό που δεν έχουμε δει είναι νομικέ ε, πρωτοβουλίε για τι ε, εργασιακέ ασθένειε. Θα ήθελα να τονίσω το, αν μιλάμε ας πούμε για την οδηγία για τη μετάθεση εργαζομένων, μιλάμε περισσότερο για την εφαρμογή, αλλά είμαστε αντίθετοι σε οποιοδήποτε είδος νέας, πρωτοβουλία, ε, νέας οδηγίας. Αν μιλάμε για ε, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή για το Ταμείο ε, για την παγκοσμιοποίηση πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά και να εξετάσουμε προγράμματα που συνάδουν με τις προτεραιότητές μας και δημιουργούν θέσεις απασχόλησης πρέπει να εξετάσουμε τις μικρομεσαίες όχι ως ένα επιπλέον ε, φόρτο, αλλά να δούμε και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τη χρηματοδότησή τους και τις σχετικές πρωτοβουλίες. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Έντιτ Χέρτζοκ για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Εμεί θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμά τη, που ήταν δύσκολο να ε, συνταχθεί, γιατί δεν υπάρχει ακόμα προπολογισμό για να το στηρίξει. Και θα ήθελα να τονίσω το γεγονό ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και διάφορα στοιχεία τα οποία δεν περιλαμβάνονται εδώ. Πρέπει να δούμε τη βιομηχανική πολιτική, αλλά να ε, καταθέσουμε και πρωτοβουλίε για την πολιτική για τι πρώτε ύλε. Θα ήταν καλό να σημειώσουμε πρόεδρο εδώ. Επάρκεια στην ενέργεια και επενδύσει στην ενέργεια. Νομίζω θα πρέπει να έχουμε πιο πολλέ απτέ πρωτοβουλίε στο πρόγραμμα τη ε, Κομισιόν. Καλωσορίζουμε το γεγονό ότι η έρευνα και η ανάπτυξη, καθώ και το σχετικό πρόγραμμα πλαίσιο, ε, θα αναπτυχθούν περισσότερο. Αν όμω αναπτύξουμε αν καταφέρουμε να φτάσουμε συμφωνία για τον προπολογισμό και για το πρόγραμμα ΙΤΕ, θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Επίσης, καλωσορίζουμε την πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί θα σημειοδοτηθεί μια επέτειος αυτής της πολιτικής σύντομα και θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένα από τα αποτελέσματα. Τους επόμενους δύο με έξι μήνες θα έχουμε προεδρία, στις επόμενες δύο εξάμεινα θα έχουμε Ουγγρική και Πολωνική Προεδρία, νέα κρατημέλη δηλαδή. Θα πρέπει να δούμε την ένταξή του. και την ολοκλήρωσή του στην Ένωση, γιατί πιστεύουμε πω το χάσμα ανάμεσα στι ανατολικέ και δυτικέ κόρε τη Ένωση, είναι απαράδεκτο, ιδιαίτερα όσον αφορά του μισθού, αλλά και άλλε πτυχέ. Θα πρέπει σε αυτά τα μέτωπα να σημειωθεί πρόοδο. Και τέλο να καλωσορίσουμε από την άποψη τη ασφάλεια σε ενέργεια τη σχετική πρωτοβουλία να γίνει κάτι, να σημειωθεί πρόοδο και για την ανατολική εταιρική σχέση. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Γκρός για 1,5 λεπτό. Δεν βρίσκεται εντό αιθούση. Περνάμε στην κυρία Κατρίν Τρότμαν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αυτό το πρόγραμμα εργασίας μιλά για ανάκαμψη της εργασίας των θέσεων ε, απασχόληση ως κλειδί για την επιστροφή στην ε, ανάπτυξη και πράγματι δεν θα πρέπει απλά να ενισχυθούν οι αποτρεπτικές ε, πτυχές που έδειξαν ότι έχουν περιορισμούς. Θα πρέπει λοιπόν η ανάκαψη να βασίζεται στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει η απασχόληση και το κοινωνικό επίπεδο να είναι δείκτες της οικονομικής ισχύω και από την πλευρά αυτή θέλω να τονίσω ότι θα πρέπει πιο σοβαρά να δούμε το θέμα του φόρου των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, να υπάρξει μεγαλύτερο συντονισμό και επίση οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Απασχόληση επίση να έχουν μια καλύτερη συνεννόηση. Σε ό,τι αφορά τώρα την απόσπαση των εργαζομένων και σε ό,τι αφορά τι υπηρεσίε γενικού ενδιαφέροντο για τι οδηγίε αυτέ πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Σε ό,τι αφορά δε την ψηφιακή ατζέντα και αυτό είναι σημαντικό ε, κομμάτι του νέου προγράμματος εργασία. διαπιστώνουμε τη φιλοδοξία της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τώρα την ηθαγένεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βάλει και πάλι τους πολίτες στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδίου. Ε, το διονοσομικό κομμάτι δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στην ασφάλεια και δει τη διαχείριση των μεταναστευτικών ε, ροών. Ολοκληρώνοντα, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι τελικά το πρόγραμμα εργασία για το 2011 θα πρέπει να είναι το παράδειγμα μια πολιτική η οποία ανταποκρίνεται θετικά σε αυτή την ε, τάση ε, ομφαλοσκόπηση που παρατηρούμε σε εθνικό επίπεδο και υποχώρηση. Έχει λοιπόν το, κοινο, το Κοινοβούλιο στο πλευρό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα στηρίξει την Επιτροπή αν δείξει περισσότερη φιλοδοξία. Grazie, σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μπροκ για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, επιτρέψατε μου να αναφερθώ σε τρία ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, θεωρώ πως στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων η Κομισιόν έχει ιδιαίτερη ευθύνη και θα πρέπει να δει περισσότερο το θέμα των ε, στρατηγικών σχέσεων αλλά και των πολυμερών σχέσεων και βεβαίως όχι από την πλευρά μόνο της ε, ε, ενέργειας ε, καθώς η στρατηγική αυτή σχέση νομίζω είναι οι στρατηγικές σχέσεις είναι προς το συμφέρον μας. Δεύτερον, δεν ξέρω τι γίνεται με τα διαρθρωτικά ταμεία και τους λοιπούς τομείς. Αλλά το θέμα της οικονομικής διαχείρισης των προγραμμάτων εξωτερικής δράσης είναι πάρα πολύ αργοκίνητο. Μέχρι να εκταμιευθούν τα λεφτά έχουν περάσει χρόνια. Και αυτό το είδαμε και στην Ανατολική εταιρική σχέση και αλλού. Ξέρω βεβαίως πως ε, έχουμε τα θέματα του προϋπολογισμού και είναι προβληματική κατάσταση όπως ήταν και πριν από 10 χρόνια με την Κομισιόν, αλλά εάν είναι να έχουν αποτέλεσμα αυτά τα λεφτά και να μην φτάνουν συνέχεια πάρα πολύ αργά, θα πρέπει να κάνουμε και μια πολιτική συμφερόντων. Οπότε θα πρέπει να βρει μια ιδέα η Κομισιόν έτσι ώστε να γίνεται πάρα πολύ γρηγορότερα η εκταμείευση των χρημάτων, να ληφθεί μια απόφαση. Και τρίτον, το θέμα του Υπερατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου και των σχέσεων με τη ΣΥΠΑ δεν νομίζω να τονίζεται αρκετά αυτή η στρατηγική σχέση στο έγγραφο της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Τον λόγο η κυρία Τικάου για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών είναι πως το 2011 θα πρέπει να εστιαστούμε στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην κοινωνική Ευρώπη. Ω αντιπρόεδρο τη Επιτροπής Μεταφορών θα ήθελα να εκφράσω την λύπη μου για το ότι αναβλήθηκε για το 2011 η Λευκή φίβλο για το μέλλον των ευρωπαϊκών μεταφορών, κάτι το οποίο είναι σημαντικό και για το μέλλον της πολιτικής συνοχής και των δημοσιονομικών προοπτικών. Όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα εργασία του 2011, θα ήθελα να τονίσω την σημασία νομοθετικών πράξεων που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τη βελτίωση της ασφάλειας ε, των δικτύων μέσω και των δημοσίων προμηθειών, της ηλεκτρονικής υπογραφής ε, και αμοιβαία αναγνώριση για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Όλα αυτά είναι απολύτω απαραίτητα για την εφαρμογή της ψηφιακής Ευρώπης και δημιουργία εσωτερικής αγοράς στις υπηρεσίες. Επίσης αναμένουμε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν τα έξυπνα ενεργειακά δίκτυα. Αυτά είναι απαραίτητα και για να εντάξουμε την ενέργεια από ΑΠΕ, στις οποίες έχουν επενδύσει τελευταία πάρα πολύ τα κράτη-μέλη, καθώς και για να δημιουργηθούν βεβαίως και υποδομές για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Καταλήγω λέγοντας πως η ψηφιακή ατζέντα και η ενεργειακή αποδοτικότητα που δημιουργούν νέες δουλειές μαζί με μια πιο κοινωνική Ευρώπη πρέπει να είναι οι βασικές προτεραιότητες για το 2011. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Δανιέλ Κασπάρη για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, έχει ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα η Κομισιόν για το 2011 και πρέπει να σας πω πως καλό θα ήταν να έχουμε πιο στοχευμένες προτεραιότητες. Έχουμε 30 γενικές διευθύνσεις, 26 επιτρόπους. Ε, δεν ανάγκη κάθε γενική διεύθυνση και κάθε επίτροπος να δικαιολογεί την ύπαρξή του με τις προτάσεις αυτές. Καλό θα ήταν για την Ευρώπη καμία φορά να έχουμε πραγματικές προτεραιότητες, να περιοριστούμε στα ουσιαστικά. Ε, δεν ε, έχει νόημα η Ευρώπη να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερα, να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στα σημαντικά. Επειδή είμαι και συντονιστή ομάδα μου στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου, θα ήθελα να φέρω κάποια πράγματα. Θα χαιρόμουν πραγματικά στι υπερατλαντικέ σχέσει, το ανέφερε ο Έλμαρ Μπροκ, επιτέλου θα σημειωθεί καμία, κάποια πρόοδο. Είναι κάθε μέρα στην ημερήσια διάταξη το θέμα, αλλά δεν υπάρχει καμία επιτυχία. Και αν βλέπετε πώ αλλάζει ο κόσμο αυτά τα χρόνια, πώ αλλάζει η οικονομική δύναμη των διαφόρων χωρών, απαιτείται ε, να συνεργαστούμε στενότερα με του Αμερικανού. Θα χαιρόμουν αν η Κομισιόν είχε πάντα κατά νου πω εδώ πέρα στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου πλέον είναι συνομοθέτης μετά τη Λισαβόνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οπότε και οι δύο πλευρέ Κομισιόν και Κοινοβούλιο, θα πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε και θα χαιρόμασταν ναι, εδώ πέρα η Κομισιόν να το λάβει αυτό υπόψη και να αφιερώσει χρόνο στον διάλογο και στην συνεργασία. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Συνάδελφε, το λόγο έχει τώρα ο κ. Μίτσελ για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον Επίτροπο που κίνησε το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κρίση να τη χειριστεί. Αλλά ο όγκος δουλειά που έχει γίνει εδώ μεταξύ και τα όσα ακόμα πρέπει να γίνουν σημαίνουν ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τον κόσμο. Εγώ είμαι συντονιστής ε, του ΕΛΚΑ στην Επιτροπή για την Ανάπτυξη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό όταν καταλαβαίνει κανείς ότι όταν συμφωνούμε να ανταποκριθούμε σε μια δέσμευση 0,07 για να βοηθήσουμε σε σχέση με το ΑΕΠ για να βοηθήσουμε τον αναπτυσσόμενο κόσμο, να σας πω ότι κάθε φορά αυτός, αυτό το κονδύλι είναι το πρώτο που κόβεται. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν το ΑΕΠ ε, μειώνεται και η συμβολή μειώνεται, η εισφορά μειώνεται, δεν πρέπει να μειώνεται ε, ανάλογα με το, η μείωση του εγχώριου προϊόντος και του εθνικού προϊόντος ε, ξανά. Ζητώ λοιπόν από την Κομισιόν μετά από την αναθεώρηση των στόχων ανάπτυξης τη χιλιετίας να εξασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη θα ανταποκριθούν στις δεσμεύσει τους. Δεν σας ζητάμε να μην, να μειώσετε τις εισφορέ, αλλά να ζητούσετε να μην μειώσουν τις εισφορέ ω ποσοστό του μειωμένου του ε, καθάριστου των χωρίου προϊόντος. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Μίτσελ και τώρα ξεκινάμε το Κατζιδιάι. Και δίνουμε το λόγο στον κύριο Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι λόγω της οικονομικής κρίσης είναι φυσιολογικό να εστιάζουμε στις οικονομικές πτυχές. Όμως η Ευρώπη δεν είναι μόνο Ευρώπη των αγορών, είναι και Ευρώπη των πολιτών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να υλοποιούμε το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης που συμφωνήσαμε να υλοποιήσουμε είναι αυτό το οποίο θα μας οδηγήσει σε μια Ευρώπη των πολιτών, συγκεκριμένα για του χρόνου. Χρειαζόμαστε περισσότερες εξελίξεις στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και γενικότερα αύξηση της ασφάλειας για τους πολίτες μας. Οι πολίτες μας ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη ασφάλεια. Θα πρέπει επίσης να ενδυναμώσουμε τον αγώνα μας κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς συγκεκριμένα. Θα πρέπει να ενισχυθούν τα δικαιώματα των πολιτών όπως επί παραδείγματι προστασία των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών και θα πρέπει να καταλήξουμε σε κοινή πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση βάση της αρχής της αλληλεγγύης. Ευχαριστώ. Κύριος Μπαλτζίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πρόγραμμα του 2011 μοιάζει αρκετά φιλόδοξο και καλό θα ήταν το έγγραφο αυτό να συνεισφέρει στο να γίνει η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πλούσια. Και στο παρελθόν βεβαίως είχαμε τέτοια φιλόδοξα προγράμματα και κάποια από αυτά δεν εφαρμόστηκαν. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά εδώ πέρα πως τα κράτη εκείνα τα οποία περνάνε σήμερα βαθιά κρίση τα θεωρούσαμε παραδείγματα οικονομικής πολιτικής αλλά μετά ήρθε η πραγματικότητα. Γι' αυτό είμαστε υπέρ της καλύτερης εποπτείας των χρηματαγορών, της ενεργειακής αποδοτικότητας και άλλων πραγμάτων. Μόνο έτσι μπορούμε να συνεισφέρουμε στο να γίνει η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και ε, να βρουν δουλειά οι άνθρωποι. Σας ευχαριστούμε κύριε, Ο λόγος του κύριο Άντριου Μπρόντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διαβάζοντα το πρόγραμμα εργασιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2011, ξεχωρίζουμε το εξή. Η χρήση τη κρίση προκειμένου να αυξηθούν ε, οι εξουσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περισσότερη εναρμόνιση δημοσιονομικών ε, και φορολογικών πολιτικών, καλύτερο συντονισμό, περισσότερη εποπτεία και φυσικά πιο ενισχυμένοι μηχανισμοί εφαρμογή. Ακούσαμε ότι έτσι θα καταλήξουμε σε υφόρο ανάπτυξη που δεν θα αποκλεί κανέναν. Το έγγραφο όμω ε, ε, της στρατηγική για το 2020 είναι πιο ειλικρινές. 23 εκατομμύρια άνεργοι, 4% μείωση του ΑΕΠ για το 2000, σε σχέση με το 2009. Δεν φαίνεται ότι ξεφεύγουμε από την κρίση. Η στρατηγική του 2020 μιλάει για τα κράτη-μέλη που είναι τα πιο καινοτόμα στον κόσμο. Βέβαια, αν οι αναδυόμενε οικονομίε κλέβουν τι εφευρέσει μα ατιμόρυτα, δεν θα μα βοηθήσει και πολύ η καινοτομία. Η στρατηγική του 2020 μιλάει για τους λόγους της Ευρώπης που είναι δημιουργικοί και ταλαντούχοι. Θα πρέπει όμως να, να ακολουθήσουμε δημογραφικές πολιτικές που θα ενισχύει αυτά τα ταλέντα και θα διαφυλάσει την δημιουργικότητά τους και την ευρηματικότητά τους. Η κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα έχει το λόγο. Ε, ε, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι φιλόδοξο. Παρ' αυτά του λείπει κάτι θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της στρατηγικής και της πολιτικής. Γιατί δημιουργούμε μια νέα στρατηγική, χαράσουμε μια νέα στρατηγική, καταρτίζουμε νέα έγγραφα. Αλλά δυστυχώς ε, πολλά θέματα, ιδιαίτερα στην ενεργειακή πολιτική, από τις προηγούμενες μας πολιτικές δεν έχουν υλοποιηθεί. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εφαρμογή. Γιατί αν δεν εξασφαλίσει την εφαρμογή των πολιτικών της ευρωπαϊκή πολιτική δεν θα διασφαλίσει την αξιοπιστία της και θα χάσει την νομιμοποίησή της. Γι' αυτό φτάσαμε και στη χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη, γιατί δεν τηρήσαμε τα κριτήρια του Μάστριχτ. Πολλέ χώρε άρχισαν να καταστρατηγούν αυτά τα κριτήρια και ειδού που φτάσαμε στα τεράστια οικονομικά προβλήματα. Ίσως δεν είναι πολύ αποτελεσματική η πολιτική. Μπορεί στα χαρτιά να μην φαίνεται πολύ ελκυστικό αυτό το θέμα τη εφαρμογή, αλλά νομίζω ότι είναι νευραλγικό σημείο για την επιτυχία μα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Λιγκεβιτσούτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Φαίνεται όμως ότι ο τομέας της απασχόλησης δεν είναι στομέα στον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει επαρκεί προτάσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω έκανε και πέρσι, παρουσιάζει τι ίδιε πρωτοβουλίε που σχετίζονται με την απόσπαση των εργαζομένων και θέλει να ρυθμίσει και τα θέματα των ε, μεταναστών εργαζομένων, αλλά αυτά δεν αρκούν. Πρέπει να σκεφτούμε και λίγο το μέλλον. Μία από τις προτάσεις ε, είναι να αυξηθεί το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Δεν παρέχεται όμως εναλλακτική μορφή ε, απασχόλησης για τους συνταξιούχους η παράνομη οικονομία αυξάνεται συνεχώς και πάλι δεν υπάρχει καμία πρόταση από πλευρά ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση του φαινομένου. Θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στην Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν να προταθεί μια οδηγία για του ελάχιστου μισθού. Ευχαριστώ το λόγο κύριο Σεκέρσκι. Ευχαριστώ. Ε, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια φαινός και από πρόταση αλλαγών αφετέρου. Έτσι έχουμε τις νέες προτάσεις για το 2011. Σίγουρα θα πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες για την ανάκαμψη την οικονομική, τη διέξοδο από την κρίση και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο για το 2011, αρκεί η στρατηγική που έχουμε εγκρίνει. Αλλά για τις αλλαγές χρειαζόμαστε ρεξικέλευθες μεταρρυθμίσεις ό,τι αφορά την οικονομική διακυβέρνηση. Έχουμε την έκθεση Μόντι που προτείνει κάποιες ε, σημαντικές λύσεις για τη βελτίωση της αγοράς. Θα πρέπει λοιπόν να προβούμε σε μεταρρυθμίσεις ε, και στην υποπτία αλλά και στη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Επίσης θα πρέπει να εφαρμόσουμε και τις λιμένες αποφάσεις ε, και να θέσουμε σε λειτουργία τις νέες υπηρεσίες και οργανισμούς. Επίσης θα πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγικότητα με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων. Βέβαια έχουμε και τις, θα έχουμε και τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές μετά το 2013 προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ε, δημοσιονομικές και οικονομικές προκλήσεις. Ευχαριστώ. Το λόγο κυρία Μόνικα Σμολκόβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Σεύσκοβιτς, είναι φιλόδοξο το πρόγραμμα εργασίας. Καλύπτει τομείς που θα μας βοηθήσουν να εφαρμόσουμε τη στρατηγική για το 2020. Πολλά υπόθηκαν ήδη σχετικά. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω πιο συγκεκριμένα πώς προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δίνει ε, στοιχεία για ταχύτερη έγκριση επιγουσών προτάσεων. Γιατί ξέρουμε πόσο ε, καιρό χρειάζεται μέχρι να υλοποιείται η ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δώσατε έμφαση στη συνεργασία Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου. Πιστεύετε όμως ότι η επικοδομητική συνεργασία με το Συμβούλιο είναι εφικτή ε, με το Σαρκοζή και τη Μέρκελ. Ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Επίτροπο κ. Σεύκοβιτς. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω ότι εκτιμώ αυτή τη συζήτηση και να ευχαριστήσω και όλα τα αξιότιμα μέλη για τα θετικά και ενθαρρυντικά τους λόγια για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι αν διατρέξουμε τις παρεμβάσεις σας μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μεγάλη σύγκληση ως προς τους στόχους που θέλετε να επιτύχουμε από κοινού και θεωρώ ότι αυτό γίνεται διότι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σε μεγάλο βαθμό κοινή απόπειρα φέτος θα θέλαμε να υπάρχει εντατικότερη επικοινωνία μεταξύ των επιτροπών. Αυτό το κάναμε και στη διάρκεια της χρονιάς και νομίζω ότι αυτό απέφερε καρπούς και εδώ έχουμε τους συλλογικούς στόχους που ε, εκπονήθηκαν από κοινού μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάποιοι από εσά ε, στάθηκαν στην κατάλληλη εφαρμογή των προτάσεων. Δεν θέλουν να παραμείνουν μόνο επί χάρτου οι προτάσεις μας. Το συμπεριλαμβάνουμε λοιπόν αυτό το αίτημα και συμπεριλάβαμε λοιπόν και στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την παρακολούθηση των εργασιών και με χαρά μου να έρχομαι σε τακτά χρονικά διαστήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σας πούμε πώς προχωρούν τα πράγματα ε, με το πρόγραμμα εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μην γίνεται συζήτηση μόνο μια φορά το χρόνο, αλλά να γνωρίζουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα πώ προοδεύουν οι εργασίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι ακριβώ κάνουμε φέτο. Μέχρι τούδε από τις 34 πρωτοβουλίες που ε, ξεκινήσαμε θα υλοποιηθούν σίγουρα οι 30. Πρόκειται για καλό στόχο εφαρμογή, αλλά βέβαια είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα και να σας ενημερώνουμε τακτικά. Επίσης χαίρομαι που μας παρακινούνται να κάνουμε περισσότερα και όχι λιγότερα, με κάποιες εξαιρέσεις, και αυτό φυσικά είναι ευπρόσδεκτο μια παρακίνηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και συμφωνώ με όλους όσους λένε ότι πρέπει να τα πάμε καλύτερα, διότι δεν πρέπει μόνο να έχουμε καλή απόδοση και να επιτυχάνουμε τους στόχους μας, αλλά να αποδεικνύουμε και ότι με υψηλή ποιότητας εργασία μπορούμε να ε, έχουμε αποτελέσματα ως καλύτερο αντεπιχείρημα για να αντιμετωπίσουμε τον ευρωσκεπτικισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αντιμετωπίσουμε τα φαντάσματα του παρελθόντος κάθε φορά που έχουμε προβλήματα προστατευτισμό, ξενοφοβία, ρατσισμό και όλα τα προβλήματα τα οποία αναφέρεται. Με καλή δουλειά και καγαστή συνεργασία μπορούμε να ε, διώξουμε τα φαντάσματα του παρελθόντος. Όσον αφορά τις υποδομές, πράγματι χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις σε υποδομές, αλλά θα πρέπει να έχουμε σύγχρονε υποδομέ για να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο και να μπορέσουμε να ε, διατηρήσουμε το ανταγωνιστικό μα πλεονέκτημα. Πρέπει να έχουμε καλύτερε υποδομέ. Αυτό δεν είναι μόνο σημαντικό για του οικονομικού μας στόχους, αλλά και για ε, πιο πράσινη οικονομία, για ε, οικονομίε οι οποίε θα είναι αποδοτικέ ω προ τι ε, τις πόρους μας και φυσικά θα πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα έχει περισσότερες επενδύσεις. Και αυτά φυσικά θα τα βρείτε στο πρόγραμμά μας. Για την ενία αγορά τώρα. Χαίρομαι για όλες τις παρατηρήσεις και για όλη την όθηση που δίνεται στην ενία αγορά, γιατί αυτό είναι το κόσμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτύχαμε πολλά με την ενία αγορά και ξέρουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε ακόμα περισσότερα εάν χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς. Πρέπει να άρουμε τους φραγμούς που εξακολουθούν να υφίστανται, πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν προσκόμματα και φυσικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τους νέους τομείς της οικονομίας. Κάποιοι από εσά αναφέρθηκαν στην ψηφιακή, ψηφιακή οικονομία. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας στην Ευρώπη αν χρησιμοποιούμε περισσότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα πρέπει να δεσμευτούμε περισσότερο σε αυτούς τους τομείς. Ο Μάριο Μόντι παρουσίασε μια εξαιρετική έκθεση. Ο Μισελ Μπαρνιέ εργάστηκε και χρησιμοποίησε αυτή την έκθεση ως βάση για το φάσμα των προτάσεών μας. Ξεκίνησε μια συζήτηση για το πώς μπορούμε να κάνουμε μια ευρωπαϊκή ενιαία αγορά καλύτερη, πιο ανταγωνιστική, η οποία θα μας φέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα για το μέλλον. Ας συμμετάσχουμε όλοι λοιπόν από κοινό, να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε το πρόγραμμα που προτείνει ο κύριος Μπαρνιέ και ποια μπορεί να είναι τα πιο επικοδομητικά για μας. Θα πρέπει να έχουμε ε, θέματα τα οποία θα αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα και έτσι μαζί από κοινού θα επιτύχουμε μια καλή νέα αγορά. Ε, γραφειοκρατικό άχθος. Γνωρίζετε ότι δίνουμε μεγάλο βάρος ε, στη μείωση του γραφειοκρατικού άχθους κατά 25% μέχρι το 2012. Να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάρα πολύ σκληρά και ελπίζουμε να το ξεπεράσουμε αυτό το όριο. Προσπαθούμε να επιτύχουμε το 30% πλέον. Θέλουμε όμως να είμαστε σαφείς. Θεωρούμε ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει μόνο από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολύ συχνά θα διαπιστώσετε ότι αυξάνεται το γραφειοκρατικό έκθος σε εθνικό επίπεδο όταν εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία με διάφορες παραμέτρους. Θα πρέπει λοιπόν να επεξεργαστούμε το θέμα αυτό από διάφορες οπτικές γωνίες και από ευρωπαϊκή σκοπιά αλλά και από εθνική σκοπιά. Όσον αφορά στην κοινωνική διάσταση της νέας αγοράς, συμφωνώ μαζί σας, μάθαμε από τα μαθήματα του παρελθόντος και θα παρουσιάσουμε ε, προτάσεις για την απόσπαση των εργαζομένων, για το χρόνο εργασίας, ε, για τις υπηρεσίες ε, κοινή ωφελία που θα δικατοπτρίζουν αυτή την πολύ σημαντική κοινωνική διάσταση. Διότι γνωρίζουμε ότι η κοινωνική διάσταση έχει αποτέλεσμα, η ενιαία αγορά συγγνώμη, έχει αποτέλεσμα όταν εναγκαλίζεται από τους ανθρώπους, από τους πολίτες και πρέπει να έχουμε ε, μια πολύ σημαντική αξιολόγηση αντικτύπου για την πρόταση που θα κάνουμε, ώστε να γνωρίζουμε ότι οι προτάσει που θα κάνουμε στους πολίτες θα γίνουν αποδεκτές και θα υποστηριχθούν από τους πολίτες. Έγινε από την κυρία Τζαβέλα μια παθιασμένη ε, αίτηση για το γεγονός ότι χάνουμε εγκεφάλους, χάνουμε τους ε, καλά καταρτισμένους ε, Ευρωπαίους που φεύγουν και πηγαίνουν να εργαστούν σε τρίτες χώρες. Ορισμένες φορές αυτό γίνεται γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν ε, φραγμοί στην αγορά εργασίας, γιατί υπάρχει έλλειψη πληροφοριών, αλλά πολλές φορές γίνεται γιατί η παιδεία δεν είναι αυτή που αναμένεται από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ε, χαίρομαι που ε, σε λίγο θα ξεκινήσει η συζήτηση για τη νέα πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Είναι εδώ και η ε, Επίτροπος Βασιλείου ε, που θα σας εξηγήσει πώς θα γίνουν τα πράγματα καλύτερα, πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις δεξιότητες και τις ανάγκες κατά τρόπον ώστε οι νέοι άνθρωποι να δώσουν νέα όθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία και να αποφοληθούμε όλοι από αυτήν. Πολλοί από εσά αναφέρθηκαν και στη σημασία του κανονισμού για τις χρηματοοικονομικές αγορές και τη σημασία ε, γρήγορης διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Πώς θέλουμε να το επιτύχουμε αυτό. Για το μέλλον ήδη επισημάναμε ότι θα θέλαμε να προχωρήσουμε με καλύτερο συντονισμό μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου και θα θέλαμε αυτό να γίνει στο πλαίσιο του νέου προγραμματισμού τη Ένωση, όπου θα αποφασίζονται ποιε θα είναι οι προτεραιότητε, ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα, ποιε θα είναι οι προθεσμίε, ώστε να έχουμε αποτελέσματα πιο γρήγορα και να επιταχύνεται η νομοθετική διαδικασία. Έτσι ε, περαιτέρω. Σας διαβεβαιώ ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από χέρι μας προκειμένου στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να γνωρίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ε, το κοινό σε εθνικό επίπεδο, τι μπορούμε να επιτύχουμε με 1% και μόνο του ΑΕΠ. Πώς είναι η δομή του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και το γεγονό ότι το 95% περίπου αυτού του προπολογισμού πηγαίνει στα κράτη-μέλη. Και αυτή η συζήτηση φυσικά θα πρέπει να περάσει και στις πρωτεύουσε. πρέπει να μιλήσουμε με τους πολίτες, να ενημερώσουμε το ευρύ κοινό για το πώς διαρθρώνεται ο προπολογισμό ώστε να έχουμε υποστήριξη για τις φιλόδοξε προτάσει μα. Ο Έλμα Μπρόκ αναφέρθηκε σε πολύ σημαντικά θέματα στι εξωτερικέ ε, σχέσει, στην ανατολική εταιρική σχέση, ε, θέματα διεύρυνσης όπου θα πρέπει να υπάρχει αξιοπιστία κατέρωθεν. Πρέπει να είμαστε και εμείς αξιόπιστοι για τον τρόπο που διαπραγματευόμαστε και παρακολουθούμε τα κριτήρια και τα πόσο πληρούνται από τα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να είμαστε και αξιόπιστοι ως προς το τι προσφέρουμε στις υποψήφιες χώρες. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι πολύ σημαντικό εταίρο και αν μπορέσουμε να άρουμε κάποιου από του φραγμού στη συνεργασία μεταξύ μα, νομίζω ότι θα είναι προ όφελό μα και νομίζω ότι θα πρέπει, ε, όπω είπε πολύ σωστά και ο κύριο Μπρόκ, να επενδύσουμε σε περισσότερη προσπάθεια για να επιτύχουμε αυτού του στόχου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί, είναι διατεθειμένη να κινηθεί, αλλά χρειαζόμαστε εταίρου. Δεν μπορούμε να έχουμε συμφωνίε τι οποίε δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει αντίστοιχη μεταχείριση και από την άλλη πλευρά. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά συνεχώς, να παρουσιάζουμε προτάσεις, να υπάρχουν ε, να βλέπουμε πού υπάρχει νέο άνοιγμα, διότι αυτό φυσικά θα είναι προς όφελος της παγκόσμιας οικονομίας και νομίζω αυτό χρειάζονται οι περισσότερες οικονομίες αυτή τη στιγμή. Τέλος, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Νομίζω ότι αυτό αναφέρθηκε πριν από λίγο. Όλοι συμφωνούμε ότι αυτό είναι ένα τομέα ε, που ενδιαφέρει και απασχολεί του περισσότερου πολίτε μα. Γι' αυτό και ακριβώ το μεγαλύτερο τμήμα του προγράμματό μα είναι αφιερωμένο στον τομέα αυτό. Οι συναδελφοί μου, κυρία Μάλστρομ και κυρία Ρέντινγκ, θα προσέξουν και θα δουν πώ μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα θέματα που ετέθησαν σε αυτή τη συζήτηση, αλλά και στο διαρθρωμένο διάλογο που έκαναν με του ε, ε ενδιαφερομένου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξεπέρασα λίγο το όριο, αλλά ήταν πολλέ ερωτήσει και προσπάθησα να απαντήσω. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο. Πέρα τη συζήτηση θα γίνει ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Διακόπτουμε για τρία λεπτά και θα περάσουμε στο επόμενο σημείο μετά. Αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Στην ε, ημερήσια διάταξη έχουμε δήλωση της Ευρωπαϊκής